αν δεν καθίστε, δεν μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Η γραπτή δήλωση που υπευλήθη από τους βουλευτές Παπαδοπούλου, Φερέιρα, Χίγκιν, Παρβανόβα και Ρωμέβα Ιρουέδα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ευαισθητοποίησης για το θέμα της καρδιακής ανακοπής συγκέντρωσε την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού μεταβιβάζεται στους παραλήπτες και θα δημοσιευθεί στα κατάλληλα κείμενα από την Ολομέλειά μας και δίνει το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους αγαπητούς συναδέλφους Jim Higgins και Αντώνια Παρβανόβα και Ρεούλε Ρωμαία Ιρουέδα και Ζωάου Φερέιρα καθώς και σε όλους τους βουλευτές που υπέγραψαν μαζί μας αυτή τη γραπτή δήλωση 11 για τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή εβδομάδα Ευαισθητοποίηση για την Καρδιακή Ανακοπή. χιλιάδε άτομα κάθε χρόνο πλήττονται από καρδιακή ανακοπή κάθε ε, χρόνο. Με ε, τις μεθόδους αντιμετώπισης αυξάνεται η επιβίωση δύο και τρεις φορές αλλά ε, μόνο σε μία από τις πέντε περιπτώσεις εξονοσοκομιακά παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια πνευμονοθερακικής αναζωογόνησης. Ε, μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά και να, χάσουμε, και να ε, σώσουμε 100.000 ζωές κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.